νέων διοριστέντων επιτρόπων εκπροσωπείται. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα σχετικά κείμενα έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις, κάποιες ενστάσεις, όχι. Έτσι τα πρακτικά εγκρίνονται, επικυρώνονται.